Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας, ε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Και αντικαθιστώ την κυρία Νικολσόνοβα. Μέχρι να έρθει, ξεκινάμε με το σημείο 17. Ευρωπαϊκό εξάμεινο, πτυχές ε, κοινωνικές ε, και απασχόλησης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ντόμπρεφ. Έχετε λοιπόν τον λόγο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Βάλτε λοιπόν τα ακουστικά. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο βασικά θέματα εδώ πέρα. Οι αυξήσεις μισθών που είδαμε τα τελευταία χρόνια δεν έχουν κάνει κάτι για τη βελτίωση των ε, μισθών, Ένα στους έξι λαμβάνει χαμηλότερο μισθό και η τάση αυτή δυστυχώς συνεχίζεται. Είναι κάτι το οποίο υποσκάπτει όχι απλά τη δημοκρατία αλλά και την ανταγωνιστικότητά μας. Βεβαίως, ε, οι κοινωνίες οι οποίες βασίζονται σε ανειδίκευτους και χαμηλόμιστους ε, εργάτες είναι καταδικασμένες ε, να καταρρεύσουν. Εμείς θέλουμε μια καινοτόμο Ευρώπη. Δεύτερον, η αντιμετώπιση της κλιματικής καταστροφής είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα αλλά βεβαίως οι πολιτικοί απαιτούν από εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους να αλλάξουν την καθημερινή τους ζωή από τη θέρμανση μέχρι το πώς δίνονται. Και έτσι θα αλλάξουν και οι επιχειρήσεις κάποιες θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν. Εάν λοιπόν δεν πάρουμε τους ανθρώπους στο πλευρό μας, Μπορούμε να έχουμε ό,τι ωραίους στόχους ε, θέλουμε, αλλά δεν θα είναι επιτυχημένοι. Εάν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ασφάλεια στη μεταβατική αυτή περίοδο, ε, δεν θα επιτύχουμε. Όταν μιλάμε για κοινωνική Ευρώπη, μιλάμε και για τις κοινωνικές πτυχές του Green Deal, για μια πιο πράσινη Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς θα τονίσω τα εξής ε, στοιχεία στην έκθεσή μου. Είναι απολύτως απαραίτητο το σύστημα φορολογίας και επιδοτήσεων των ε, κρατών μελών να μειώσει τις εισοδηματικές ε, διαφορές. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται μια συνολική στρατηγική κατά της ε, φτώχειας, της παιδικής φτώχειας. γιατί ήδη από τα σχολεία ξεκινάει η κατάσταση αυτή, γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε στο σύστημα της εκπαίδευσης και στην καταπολέμηση της φτώχειας. Μόνο έτσι θα μπορέσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν στο και χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα εγγύησης για τα παιδιά. Μετά, η θέση των ε, γυναικών. Πρέπει να βελτιωθεί. Έχουμε κάνει πολλά, αλλά δεν αρκούν. Και έχουμε συνεχώς ε, νέες προκλήσεις που ανακύπτουν. Η απασχόληση των νέων γυναικών. Γυναικών που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας ε, έχουν ειδικά προβλήματα και νέες ε, προκλήσεις. Οι γυναίκες ε, που ασχολούνται με την οικογένεια, με τους άρρωστους ή τους ηλικιωμένους. Και αυτές πρέπει να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Η εμπειρία τους είναι απολύτως απαραίτητη. Πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες για όλες αυτές. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε λοιπόν το θέμα των παιδικών σταθμών και τα στοιχεία κοινωνικής πρόνοιας. Κάτι άλλο. Η οικονομία τα επόμενα χρόνια πιθανότατα θα επιβραδυνθεί. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψει την προσοχή των θεσμικών οργάνων στις ε, συνέπειες ε, και τις εμπειρίες ε, της διαχείρισης της κρίσης 2008-2019 ε, είδαμε ότι οι κοινωνικές δαπάνες δεν μπορούν να περικοπούν. Είδαμε τι επιπτώσεις έχει αυτό. και πώς επηρεάζει την ε, ειρήνη, την κοινωνική. Και από τις ε, διάφορες κοινωνικές πτυχές ε, βλέπουμε ότι πρέπει αυτά να είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχει πράσινη Ευρώπη, ισχυρή Ευρώπη χωρίς κοινωνική Ευρώπη. Αυτά ήθελα να τονίσω στην έκθεσή μου. Λοιπόν, τροπολογίες μέχρι τις 28 Ιανουαρίου, στα αγγλικά γιατί ο χρόνος πιέζει και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει το ισχυρό μήνυμα. Να ενισχυθεί δηλαδή, όχι απλώς να διατηρηθεί η κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ναι, εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσή σας. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα πάρουν πρώτο το λόγο οι συντονιστές. Ο κύριος Ράτκε πρώτος, παρακαλώ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σας και τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Και σας ευχαριστώ για την εντατική προεργασία και την ανταλλαγή απόψεων που ήδη είχατε με κάποιους ε, σκιώδεις ηγητές και την επιζητήσατε τη συνεργασία. Σε σχέση με αυτά που άκουσα τώρα, και σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε, μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποια που πηγαίνουν σωστή κατεύθυνση. Καλά, θα διαπληκτιστούμε και για κάποιες λεπτομέρειες, αλίμονο. Γι' αυτό έχουμε προγραμματίσει και συνεδρίαση των σκιωδών. Και χαίρομαι ε, για την κοινή μας προσπάθεια και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον. Ευχαριστώ, κυρία Γιον Κέριος. Θα είμαι σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω την Κλάρα, τη συνάδελφό μου, ε, για την παρουσίαση της έκθεση και για την εκπόνηση, γιατί έχει δουλέψει σκληρά. Αφήστε δε που έπεσε και χριστουγεννιάτικα αυτή η δουλειά της έκθεσης και πιέζει και ο χρόνος. Οπότε, ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Εγώ δεν έχω πάρα πολλά σχόλια να κάνω επί του περιεχομένου. Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου μπορεί κάτι να σκεφτώ και να κάνω και καμία τροπολογία. Θα τα δούμε αυτά στη συνεδρίαση με τους κοιόδης ηγητές. In a good way. Yes, thank you very much, Madam. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βαντρέν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, λέει κυρία Βεντρέν, για το έργο της και την εργασία της είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εμείς χαιρόμαστε ε, από την πρόθεση και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βάλει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τον κοινωνικό πυλώνα. Και η στρατηγική που προτείνει επίση η ετήσια εγγράφεται σε ένα αβέβαιο οικονομικά πλαίσιο όπου η κοινωνική διάσταση δεν θα πρέπει να παραμεληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβε πόσο επίγον είναι το θέμα και ενέγραψε σε μια ευρύτερη στρατηγική το Πράσινο Σύμφωνο όλα αυτά τα θέματα. Μια οικονομία χωρίς άνθρακα θα πετύχει μόνο εάν είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και δεν παραμελήσει κανέναν. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ουσιαστικά μέτρα να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους εργαζόμενους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για βιώσιμες θέσεις εργασίας με χρηματοδότηση της ε, μετεκπαίδευσης και του μετασχηματισμού της οικονομίας. Και γενικότερα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν τις συστάσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η πρόεδρος διακόπτη. Μήπως να διαβάζετε λίγο πιο αργά για να σα προλαβαίνουμε. δεν αρκεί να πλαισιώσουμε και να βοηθήσουμε την οικολογική μετάβαση. Χρειάζεται να χτίσουμε την κοινωνική Ευρώπη, όπως τονίζει η στρατηγική αιτήσια της ε- Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ψηφιοποίηση έχει επιπτώσει στην εργασία. Μπορεί να φέρνει ε, τον κόσμο που δεν έχει δουλειά ε, στην αγορά εργασίας, αλλά υπάρχουν νέε προκλήσεις και προβλήματα που οι εργαζόμενοι σε επιγραμμικές πλατφόρμες που έχουν πρόβλημα γιατί δεν είναι ασφαλισμένοι. Κινδυνεύει επίσης με την ψηφιοποίηση κάπως να επιβραδεθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Θύμησε η συγκήτρια πόσοι ε, απειλούνται από τη φτώχεια, ιδιαίτερα γυναίκες, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Αφήστε δε, ε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού και επισφάλειας πολύ μεγάλης ένδυας. Αυτό ε, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με μέτρα υπέρ των νέων, με την εγγύηση για την νεολαία ή με την εγγύηση για ε, τα παιδιά, για να μην υπάρχει παιδική φτώχεια. Καταπολέμηση λοιπόν της φτώχειας, ενίσχυση της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας των νέων πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Και θα πρέπει να φροντίσουμε, να επαγρυπνούμε, να παραμείνει η χρηματοδότηση στα επίπεδα που πρέπει. Είναι η πρώτη φάση τώρα διαβούλευσης με τους κοινωνικούς ε, εταίρους για ένα ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, ένα κατώτατο μισθό βέβαια σε κάθε χώρα ε, που να εγγυάται την κοινωνική σύγκληση προς τα πάνω. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, ε, κύριος Ντομπρόφσκης, έχει ως τίτλο του χαρτοφυλακίου του «Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων». Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έτσι ώστε να είναι πραγματικό εργαλείο στην υπηρεσία της κοινωνικής Ευρώπης ε, που να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ψηφιακής και της κλιματικής εποχής ε, και αλλαγής. Η κυρία Λάγκεν Ζήμπερ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Πρασίνων θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κλάρα Ντόμπρεφ για την ε, καλή δουλειά που έκανε Καλωσορίζω την εστίαση που δίνει το σχέδιο της έκθεσης. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ένα πλαίσιο για το κατώτατο εισόδημα, όπως είπαν οι συνάδελφοι, και να ε, κλείσει η ψαλίδα των φύλων, η μισθολογική. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προετοιμάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να εκπονήσουν στρατηγικές ε, που να, για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης. Εκεί βοηθούν και κάποιες ΜΚΟ που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. Έχουμε ε, καταρτήσει και τροπολογίες για θέματα στέγασης και αναπηρίας. Αυτά. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ και περιμένω τη συνεδρίαση των σχεδόν. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, σας ευχαριστώ και εγώ για την έκθεση. Έχετε ξεκινήσει με αφετηρία το ότι το πράσινο deal θα οδηγήσει σε ανάπτυξη και ευημερία. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει το αντίθετο. Καταστρέφει χιλιάδες καλές θέσεις εργασίας. Δεν μιλάμε μόνο για άνθρακα, μιλάμε και για το χάλιβα και την αυτοκινητοβιομηχανία. Μόνο στην ε, Γερμανία μιλάμε για 400.000 θέσεις εργασίας που απειλούνται. Και βεβαίω ε, μιλάμε για τον Χάλβα. Εδώ πέρα δηλαδή, αν κόψουμε τις ρίζες ενός δέντρου, το δέντρο θα πεθάνει. Η Αγγλία δεν μας εγκαταλείπει, δεν μας χωρίς λόγο. Ε, κοιτάξτε και το εξή. Ε, μιλήστε για του άστεγου, οι οποίοι αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκτό από τη Φιλανδία που έχει την λύση με το πρόγραμμα Housing First. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αυξάνονται τα νίκια. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αυξηθεί κατά πάνω από 50%. Γιατί. Ε, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η πολιτική των αρνητικών επιτοκίων έχει συνεισφέρει ε, στο να επενδύει ο κόσμος στον πετόν. Γι' αυτό ανεβαίνουν τα ακίνητα. Μετά έχουμε μετανάστες, παράνομους μετανάστες. Κάπου πρέπει να μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όσο περισσότεροι μπαίνουν στην ε, αγορά και να ζητούν στέγη, ανεβαίνουν τα νίκια. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Και θεωρώ ότι στα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, εδώ πέρα φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κυρία Φόλσκα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Είναι σαφής, ε, κάτι το οποίο δεν σημαίνει πάντα. Ε, υπάρχουν κάποιοι τομείς που είναι σημαντικοί. Η άστεγοι, άνθρωποι που έχουν περιθωριοποιηθεί, ζητήματα κοινωνικής ανισότητας, ε, τα παιδιά, η κατάσταση στην αγορά εργασίας ε, και η ανεργία. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν, αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι όταν η ανάπτυξη είναι καλύτερη, οι επενδύσεις ε, κατευθύνονται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Αν μιλάμε για ανάγκες, εννοούμε την εγγύηση για τα παιδιά, τον βασικό μισθό και αναμένουμε να μάθουμε ποιες ε, θα είναι οι λύσεις που θα δοθούν. Γιατί όλα αυτά ακούγονται κάπως ε, γενικά λέμε ότι δεν πρέπει να μειωθεί η χρηματοδότηση της πολιτικής ε, συνοχής. Μιλάμε για το ταμείο, το κοινωνικό. Και εδώ πέρα θέλω να συμφωνήσω με τον ε, συνάδελφο για τον Green Deal. Πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική Ευρώπη. Γι' αυτό το ερώτημα είναι εάν σκέφτεται καθόλου και τους εργαζόμενους η Ευρώπη τους εργαζόμενους που δεν θα έχουν νέες θέσεις εργασίας οπωσδήποτε αλλά αυτούς που θα χάσουν τη δουλειά τους. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί κανείς δεν θα περιέγραφε μια τέτοια μετάβαση ως δίκαιη. Επίσης ε, αναφέρονται τόσα πολλά κοινωνικά προβλήματα εδώ πέρα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να λυθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Η συναρφός δεν είναι εδώ. Οπότε αυτά. Κύριε Κώσα. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή είναι μια ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την εγκρίνουμε κάθε χρόνο και παρακολουθούμε το θέμα αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα γίνονται πολλές τροπολογίες ε, και αυτό δείχνει ε, πόσο ενδιαφέρεται το Κοινοβούλιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που συζητούμε την έκθεση αυτή και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία μας ε, στο προσεχές μέλλον. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, πολύ σημαντικό, θα έρθουν πάρα πολλέ τροπολογίες. Επιτρέψτε μου να τονίσω τα εξή ε, στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ναι, είναι ισορροπημένη η έκθεση. Ξέρω ότι οι ομάδες θα διχαστούν για τα διάφορα θέματα ουσίας. Όσοι συνάδελφοι είναι παρόντες, ε, θα κάνουν τροπολογίες έχουν τον ίδιο στόχο. Όλοι μας θέλουμε μια πραγματική κοινωνική Ευρώπη με κοινωνικές λύσεις για τα προβλήματα. Όλοι στην Επιτροπή Απασχόλησης έχουμε αυτό το στόχο. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν ρόλο τα κράτη-μέλη εδώ και θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις προτάσεις που θα κάνουμε έχω προτάσεις για λύσεις και ελπίζω να τις λάβετε υπόψη και να τις συμπεριλάβετε στο κείμενο. Συμφωνώ πάρα πολύ ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ένα εργαλείο για την ε, οικονομική αλλά και την κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω όμως να προειδοποιήσω για κάτι μην την παραφορτώσουμε αυτή τη βάρκα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικές απαιτήσει. Ναι, δεν λέω να προσθεθούν και άλλα θέματα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά το σημαντικότερο ε, όλων είναι να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, Θυμάστε στις ακροάσεις των επιτρόπων, τους είχαμε ρωτήσει. Ο κύριος Δομπρόφσκης είπε ότι δεν πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να είναι λύση. Ένας κατώτατος μισθός πανευρωπαϊκά. Εδώ καλά καλά υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν ε, έχουν εγγυημένο κατώτατο μισθό. Στο Λουξεμβούργο είναι 2.200 ευρώ, Α πούμε, στη Βουλγαρία είναι 200 ευρώ κατώτατο μισθό. Εγώ θα πρότεινα να βρούμε μια άλλη λύση. Να προσπαθήσουμε από κοινού να ορίσουμε ένα πλαίσιο μαζί με τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν τέτοιες τεράστιες διαφορές. Επίσης, υπάρχουν πολλά έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν για τη μετάβαση. Και έχουμε προβλέψει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Δεν θα πρέπει όμως να πάρουμε κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση αυτή αν μπούμε σε ένα τέτοιο δρόμο. Συμφωνώ με την εισηγήτρια και την υποστηρίζω. Είμαι βέβαιος ότι θα τονίσει και η συγγήτρια ότι δεν υποστηρίζουμε τα βήματα εκείνα που αποδυναμώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και επίση χαίρομαι που αναφέρετε τα άτομα με αναπηρίε γιατί χρειάζονται την υποστήριξή μα. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Θέλω να σα θυμίσω λίγο το χρονοδιάγραμμα. Ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 28 Ιανουαρίου, έγκριση στην Επιτροπή μας στις 20 Φεβρουαρίου. Uh, Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Ντόμπερ. Όχι, προσβλέπω στη συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για να έχουμε τελικά μια ισχυρή έκθεση και δίκαιη έκθεση. Περνάμε στο 18 τώρα. ενισχυμένη συνεργασία. Κανονικά η συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει στις 3.30. Φοβάμαι ότι δεν είμαστε όλοι παρόντες και παρούσες. Θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον να έρθει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο εισηγητής φυσικά. Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. sorry everyone for waiting. We will uh, for certain points in the... Λοιπόν, είπαμε ότι είναι ενδεικτικό ε, το χρονοδιάγραμμα που βάζουμε για τις συζητήσεις, αλλά δεν γίνεται δουλειά έτσι και φοβάμαι ότι θα πρέπει να περιμένουμε δεν έχουμε όλους τους σκιώδεις, ήρθε ο συγητής, δεν είναι πάρα πολύ άδικο. Ε, κάνουμε τη συζήτηση ερήμην τους, άρα πρέπει να περιμένουμε λίγα λεπτά. περιπτώσεις. Okay, dear colleagues, it looks like we are complete now. Uh, thank you, especially to... Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ιδιαίτερα τον εισηγητή που ήρθε νωρίτερα. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις εργασίες μας. Αυτό με τα, τις χρονοθυρίδες δεν λειτουργεί και μπορούμε να το βελτιώσουμε πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε λοιπόν στο σημείο 18 ε, το σχέδιο έκθεσης για ε, την ενισχυμένη συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πισάρο. Θα μιλήσω την Πορτογαλική. Με μεγάλη ικανοποίηση ανέλαβα τη συγκεκριμένη θεματολογία τα θέματα των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο στόχος της πλήρους απασχόλησης που είναι σημαντικό βήμα κοινωνικής προόδου ε, διαπνέει θα έλεγα τις βασικές αρχές, τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς λοιπόν το θέμα είναι να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στις υπηρεσίες απασχόλησης των διαφορετικών κρατών μελών. Θα πρέπει όλοι μας στο σύνολο ε, να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε τις χρήσιμες εμπειρίες σε κάθε χώρα στον τομέα της ε, γνωστοποίησης ε, και ανταλλαγής πληροφοριών. Νομίζω ότι η πρόταση συνεπώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια χρήσιμη πρόταση και ε, διακρίνω αρκετά πλεονεκτήματα Διαπιστώνω επίσης με ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάποιες αναφορές στη λεγόμενη βάση ε, στην έδρα των κοινωνικών δικαιωμάτων και στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε κάποιες πλευρές, ε, ε, κάποιες μέσω των τροπολογιών, ε, γύρω από τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε. Η στρατηγική 2020 έτσι όπως περιγράφεται νομίζω έχει ξεπεραστεί. Θα πρέπει να επανέλθουμε στον στόχο για την πλήρη απασχόληση και συν της άλλης θυμίζω ότι αυτά αναφέρονται στα άρθρα 3 και 9. Ήδη έχουμε επανέλθει ότι τα λεγόμενα benchmark θα πρέπει να καθοριστούν εκ νέου με βάση το άρθρο 11 και εδώ εντάσσεται η προβληματική για τους μακροχρόνια ανέργους όπως επίσης και για αυτούς οι οποίοι έχουν θέματα αναπηρίας. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών και αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα με τον συντονισμό μεταξύ τους. και φυσικά θα πρέπει για να γίνει αυτό να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές οι οποίες έχουν επισυμβεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας. Και αναμένουμε ακόμα περισσότερες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Αυτό που είναι προφανές είναι ότι θα πρέπει να αναδιαμορφώσουμε τις ε, υπηρεσίες απασχόλησης. Είναι επίσης σαφές ότι πέρα από την αμοιβαία αν θέλετε ενημέρωση να ανταποκριθούμε με πολύ πιο συγκεκριμένο από ό,τι σήμερα τρόπο ε, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίος πολίτης, δηλαδή ε, ανεργία των νέων, προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανανέωση της ισχύω του δικτύου αυτού για 7 ακόμα χρόνια και είναι μια πρόταση θετική και θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να θεσμοποιήσουμε καλύτερα το δίκτυο αυτό, αλλά παρόλα αυτά η προθεσμία αυτή δίνει τη δυνατότητα και συλλογή στοιχείων και ε, τακτοποίησης, ταξινόμησης μάλλον των στοιχείων αυτών και στη συνέχεια αξιολόγησής τους. Προβλέπετε λοιπόν κάτι τέτοιο. Το θέμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και να είναι προσυζήτηση και για μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θα κατατεθούν και άλλες τροπολογίες και ελπίζω τελικά να έχουμε μια καλή έκθεση η οποία θα μας δείξει πόσο θετική είναι η πρωτοβουλία αυτή, η οποία εκλαμβάνεται πάρα πολύ θετικά από όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Μια ανταλλαγή απόψεων τώρα των ε, σκιωδών εισηγητών. Ξεκινάμε την κυρία Σκητέλα. Σας ευχαριστώ αγαπητέ κυρία, λέει η κυρία Σκίτενταλ. Το δίκτυο αυτό έχει αποδειχθεί μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και βοηθάει τους ε, πολίτες να βρουν μια καλή δουλειά. Αποτελεί λοιπόν ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσθέσει αξία όσον αφορά την αγορά εργασίας. Ε, συνεισφέρει στον εξυγχρονισμό και ενίσχυση σε δημόσιες ε, υπηρεσίες έβρεση εργασίας. Αυτό γίνεται μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και της ανταλλαγής ε, βέλτιστων πρακτικών. Θα θέλαμε λοιπόν ε, το ΕΛΚ να δει μια περαιτέρω συνεργασία. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο βελτιώσεων, όμως το μεγαλύτερο ζήτημα τα επόμενα χρόνια είναι ο κόσμος εργασίας που αλλάζει. Η αγορά εργασίας θα διαταραχτεί λόγω ψηφιοποίησης και παγκοσμιοποίησης και την ανάγκη επανεκπαίδευσης. Αναφέρατε ήδη κάποια από αυτά τα ζητήματα, όμως από την ε, σκοπιά του ΕΛΚ θα θέλαμε να τονίσουμε αυτά τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η ανάγκη κατάρτισης, ψηφιοποίηση, επίσης προσφορά και ζήτηση και τέλος η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες απασχόλησης. Τέλος, είναι ένα σχέδιο έκθεση, είναι πάρα πολύ καλό νομίζω και αναμένω την ε, περαιτέρω συνεργασία μας ε, για να καταλήξουμε σε κάποια πολύ θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Βελή. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω την ε, βουλγαρική. Κυρία η κύριε Πιτσάρο συμφωνώ πως ε, οι ευρωπαϊκές ε, υπηρεσίες αυτές θα ενισχύσουν ε, τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης στον τομέα της διοίκησης καλοδεχόμενη πρόταση της εισηγήτριας να εστιάσουμε στις ανάγκες για μια πιο έντονη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών εταίρων και να δούμε και τις υπηρεσίες ε, ξέβρεσης εργασίας και θα πω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και των άλλων παρόχων ε, κοινωνικών υπηρεσιών για να διευκολύνουμε αυτούς που αναζητούν εργασία. Ε, θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε ε, με το να βελτιώσουμε το περιβάλλον ε, λειτουργίας τους, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Θεωρώ ότι οι δημόσιες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο των ε, εργαλείων αυτών. Παραδείγματος χάρη ε, βάσεις δεδομένων που αποτελούν ε, τον δεσμό μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Θα πρέπει λοιπόν να στηριχθούν στο εθνικό επίπεδο για να απτυχθεί η απαραίτητη αυτή ικανότητα μέσω του κατάλληλου προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού. Επίσης είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα ε, μέσα να με, και τα μέσα μέτρησης ε, των αποτελεσμάτων των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης ε, να φροντίσουμε οι υπηρεσίες αυτές να είναι αποτελεσματικές όμως δεν στηρίζω την πρόταση που περιέχεται στην τροπολογία 14. Αναφέρονται εκεί πέρα διάφορες ε, ευπαθείς ομάδες, αλλά δεν αναφέρονται οι νέοι από ομάδες ή οι πρόσφυγες και μετανάστες. Λοιπόν, εδώ πέρα μπαίνουν οι βάσεις ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της ανάπτυξης ε, ο κύριος Σατουρή, ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω ε, πραγματικά να επενέσω το ε, έργο του εισηγητή και να τον ευχαριστήσω γιατί έκανε προσπάθεια να συμπεριλάβει τις προτάσεις μας ε, στο σχέδιο έκθεση. Χαίρομαι που αναφέρεστε στην ισότητα των φύλων στην αξιοπρεπή ζωή και, τη, και εργασία και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Όλα αυτά τα υποστηρίζω και εγώ και θα μπορούσε αυτό να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Η πολιτική μου ομάδα ε, θέλει να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή και κυρίως τα εξή. Θέλουμε να προτείνουμε το δίκτυο ε, να μην έχει χρονικό περιορισμό μέχρι φυσικά ε, να ληφθεί απόφαση που θα ορίζει διαφορετικά ε, μια απόφαση που μπορεί να έρθει ανα πάσα στιγμή. Εμείς δεν θέλουμε να παγιώσουμε, ε, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο θεσμό, αλλά να συνεχιστεί ε, καλή πρακτική και να αξιολογείται και η υπεραξία κάθε πέντε χρόνια. Δεν είναι λευκό επιταγή, ούτε τίποτα κατοχυρώνεται έτσι στον αιώνα τον άπαντα, αλλά ε, συνεχίζουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, της συνεργασίας των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Επίσης, ε, θέλουμε να τονίσουμε την ποιότητα της βοήθειας που παρέχεται. Πολλές φορές οι άνεργοι έχουν προβλήματα λόγω του ψηφιακού χάρματος, λόγω της φτωχοποίησης των νέων που δεν βρίσκουν δουλειά, που δεν έχουν αρκετή εκπαίδευση, κατάρτιση, μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι αποκλείονται από την αγορά εργασίας και από την κοινωνία πολλής και, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θέλουμε λοιπόν να δίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια ε, να γίνεται μάλλον ιδιαίτερη προσπάθεια για να υπάρχει ατομική πλαισίωση, βοήθεια. Είναι τόσο περίπλοκες οι καταστάσεις και τόσο διαφορετικές που πρέπει και το προσωπικό να μετακπαιδεύεται, το προσωπικό ε, των υπηρεσιών ε, απασχόλησης που είναι ε, η πρώτη στους οποίους απευθύνεται κάποιος για να βρει δουλειά, ε, έτσι ώστε να μπορούν να βοηθούν όσο γίνεται καλύτερα και ε, στοχευμένα. Επίσης, Θέλουμε να ασχοληθούμε και με τα νέα επαγγέλματα, πράσινα επαγγέλματα. Ποια είναι αυτά για να μετασχηματιστεί η οικονομία μας. Εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδέσουμε τη δουλειά που κάνουν οι ε, ε, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης με τους στόχους της νέας πράσινης συμφωνίας. Και αυτό θέλουμε να διαπερνά ε, ολόκληρη την αυριανή ευρωπαϊκή κοινωνία. Δίκαιη και κοινωνική μετάβαση σημαίνει και πλαισίωση και καλύτερες δεξιότητες και προσόντα των ανέργων έτσι ώστε να βρουν καλή δουλειά. Ε, ευχαριστώ η κυρία Ζαμπέλη. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Διάβασα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνώ με την παράταση της ενισχυμένης συνεργασίας και υπό το φως των στατιστικών που έχουμε πάρει από το Κέντρο Μελετών έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το μέσο αυτό, να λειτουργήσουμε το, το μέτρο αυτό ε, με πιο ικανοποιητικό τρόπο. Ritengo tuttavia che il lavoro da fare da qui Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν μέχρι το 2017, αλλάζοντας εντελώς την ομοθεσία για την απασχόληση, γιατί μέχρι τώρα δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σωστά. Προχωρά επίσης και η ψηφιοποίηση ε, των, της, των θέσεων εργασίας σε γραφεία και να συνεχιστεί η λειτουργία του ε, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η ανταλλαγή επίσης ε, εμπειριών ανάμεσα στις υπηρεσίες απασχόλησης είναι απαραίτητη έτσι ώστε εκεί όπου τα πράγματα πηγαίνουν καλά να μπορέσουν να ενημερώσουν σωστά και τις υπέλοιπες χώρες οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια περαιτέρω θέματα. Η κυρία Ραφάλσκα θα μιλήσει εξ ονόματος ε, της σκιώδης συγγήτρια από την ομάδα της. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της ομάδας των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, υποστηρίζουμε το αίτημα επίσημης συνεργασίας των ε, διαφόρων εθνικών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Πραγματικά να δημιουργηθεί ένα τέτοιο άτυπο δίκτυο, αυτό βοήθησε για την καταπολέμηση της ανεργίας έγινε πιο ομαλή η συνεργασία των οργανισμών στα κράτη-μέλη και ήταν και αμοιβαία υποφελής, γιατί με τη σύγκριση ο καθένας διδάσκεται από τον άλλον. Ε, και θα ήταν σκόπιμο να ε, παραταθεί ε, μέχρι τις 31 Δοδεκάτου του 2027 για μια επταετία αυτή η συνεργασία δηλαδή να ανανεωθεί. Είναι πολύ σημαντικό οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης να συνεννοούνται, ε, να συνεργάζονται, γιατί έτσι αυξάνεται και η ίδια αποτελεσματικότητα. Αυτό υποστηρίζεται με διάφορα μέσα και εργαλεία που υπάρχουν. Ε, υπάρχει αυτοξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, ε, θεματική αξιολόγηση, ας πούμε δεξιότητες και ακόμα και η ποιότητα το, της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ε, διοργανώνουν διάφορες ημερίδες, την Ευρωπαϊκή ημέρα εργαζομένων, εργοδότη. Ε, γενικά είναι καλά τα εργαλεία για την υποστήριξη της δουλειάς που κάνουν αυτοί οι οργανισμοί απασχόλησης. Καλό είναι να συνεννοούνται υπηρεσίες, γιατί ε, έτσι προωθείται η Ευρώπη που μας ενδιαφέρει. Έχει κάποιες πρωτοβουλίες αυτό το δίκτυο που θα πρέπει να βοηθούν για να βελτιώνονται οι εθνικοί οργανισμοί. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, συμφωνούμε με τις περισσότερες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν επιφυλάξεις ε, ως προς τη διατύπωση ορισμένων τροπολογίων. Εγώ έχω αντίρρηση με τη διατύπωση που λέει ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και με τρίτες χώρες. Καλά, η συνεργασία δεν βλάπτει. Καλό είναι να έχουμε επαφές ε, και έχει ωφέλη και επιτυχίες. Αλλά αυτό να μπορεί να το αποφασίζει το κάθε κράτος μόνο του, αν θέλει να συνεργάζεται με τρίτη χώρα. Με τον εκάστοτε, ο ΑΕΔ, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να επιβληθεί με κάποιο νομοθέτημα. Θα κάνουμε και εμείς τροπολογίες και θα τις υποβάλουμε εγκαίρως. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο σκιώδης εισηγητής της ΓΚΟΕ είναι άρρωστος. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για τροπολογίες είναι η 30 Ιανουαρίου. και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας είναι 26 Μαρτίου. Κύριε Ισηγητά, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια σχόλια μόνο για τα όσα ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν πρέπει ε, να σκεφτόμαστε ότι το δίκτυο αυτό θα αλλάξει τις υπηρεσίες της χώρας. Αυτό το κάνει κάθε χώρα μόνη της. Δεν θα υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή διοίκηση των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ε, υπάγονται στην κάθε χώρα. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να δημιουργήσουμε ένα μέσο για να επιταχυνθεί η αλλαγή. Ε, και ακριβώ αυτό είναι ο στόχο, να δεχτούμε ένα από τον άλλον από τι εμπειρίε ε, θετικέ, αρνητικέ. Έχω μιλήσει με πολλού ανθρώπου Και ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος για δουλειά που έχει κάνει. Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου μπορούν έτσι να απαντήσουν καλύτερα σε κάποια ζητήματα, π.χ. στα θέματα προσφύγων και μεταναστών που ανέφερε μια συνάδελφος, η απάντηση ήταν ευκολότερη γιατί οι υπηρεσίε έμαθαν η μία από την άλλη πώς να αντιμετωπίζουν διαφορετικούς πολιτισμούς και διάφορα ζητήματα. Έχουμε βεβαίως την δυνατότητα να επιφέρουμε ακόμη περισσότερες αλλαγές και ε, θα τις ε, τροπολογίες σας. Υπάρχει συζήτηση. Η εξής, να το παρατείνουμε για 7 χρόνια ή να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο σύστημα. Το Κοινοβούλιο καλό είναι να λάβει μια απόφαση για 7 χρόνια. Θα μας δώσει έτσι περισσότερη δύναμη να παρέμουμε στη συζήτηση αυτή. Και αυτή είναι η απόφαση που θα ικανοποιήσει και τις υπηρεσίες. Γιατί ξέρουν ότι έτσι το Κοινοβούλιο θα τους ξαναφωνάξει να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορούμε να, να στείλουμε ως πολιτικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ και περνάμε άρα στην παρουσίαση ε, τριών πράξεων κατεξοδότηση από την ε, Κομισιόν θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Μέρση που ήρθε από το Λουξεμβούργο να έρθει εδώ πέρα σήμερα και βεβαίως ε, θεωρώ ότι τα αξιόπιστα δεδομένα και δείκτες ε, είναι ο πυρήνας χάραξης σωστής πολιτικής, ειδικά στην κοινωνική πολιτική, για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια για να στοχεύσουμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να βρούμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία των πολιτικών μας. Χρειαζόμαστε δεδομένα. Οπότε θα ήθελα να σας δώσω τον λόγο κύριε Μέρση για να συζητήσουμε τις πράξεις ε, κατεξιοδότηση για το πολιετές ε, πρόγραμμα που τίτλο έχει τον αριθμό και τον τίτλο των μεταβλητών για την ε, έρευνα της αγοράς εργασίας, του εισοδήματος και των συνθήκων ζωής. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο αλλά και τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή που συνεργάστηκαν ε, για να επιτύχουμε αυτή την απόφαση στον κανονισμό πλαίσιο κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή για τις ε, τρεις πράξεις εξοδότηση. γιατί σχετίζονται στενά και οι λόγοι είναι παρόμοιοι. Ο βασικός κανονισμός που, που λέγαμε yes, δηλαδή ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές ε, κοινωνικές ε, στρατηγικές ε, και θέλαμε ακριβώς να δώσουμε αυτό το θετικό μήνυμα. Εγκρίθηκε το 2019 από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αφορά τα βασικά στατιστικά στοιχεία για τα κοινωνικά θέματα. Καλύπτει δηλαδή κάποια βασικά ζητήματα που είναι καθημερινά στις εφημερίδες. Απασχόληση, φτώχεια, υγεία. Ναι, ζητήματα θεμελιώδη για τα κοινωνικά στατιστικά στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά αυτού του κανονισμού είναι ότι οι πληροφορίες συλλέγονται από τα νοικοκυριά και τα άτομα. Δεν είναι στατιστικά δεδομένα, είναι πληροφορίες για τα άτομα και τα νοικοκυριά. Μας δίνει ένα ενιαίο πλαίσιο από πολλές ε, διάφορες έρευνες, ε, δηλαδή την έρευνα για την αγορά εργασίας, ε, την έρευνα για το εισόδημα και τις συνθήκες ζωής, την έρευνα κατανάλωσης, την έρευνα για την υγεία, την εκπαίδευση, χρήση πληροφορικής από τα νοικοκυριά και την έρευνα χρήσης ε, χρόνου. Για πρώτη φορά λοιπόν όλα αυτά τα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα ένας κανονισμός. Γιατί έχει υποβάλει το νέο κανονισμό η Κομισιόν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι μελέτες αυτές σχεδιάστηκαν ε, σταδιακά καθώς εμφανίζονταν οι ανάγκες ε, τη δεκαετία του 1990 και προσαρμόστηκαν στην κατάσταση και στις ανάγκες που υπήρχαν τότε αλλά αντιδρούσαν μόνο με βάση το πώς είχαν οικοδομηθεί. Επίσης είχαμε νέες ε, ανάγκες, νέες απαιτήσει από τα δεδομένα αυτά Παραδείγματο χάρη να έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπου έχουμε ένα πίνακα βαθμολογίας που βασίζεται κατά 80-90% στις έρευνες αυτές. αυτό το οποίο λέμε η οικονομία η οποία λειτουργεί για τους ανθρώπους, ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, που αφορούν την κοινωνική διάσταση και διάφορους πίνακες βαθμολογίας για τα κοινωνικά της Κομισιόν. Ο κανονισμός αυτός έχει στόχο τον βάλει όλα αυτά τα δεδομένα σε ένα πλαίσιο για λόγους πολιτικής αλλά και διάφορους τεχνικούς λόγους τώρα δεν θα αναφερθώ. Αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες κατηγορίες ανθρώπους σε όλο το φάσμα συλλογής πληροφοριών και όχι ε, μεμονωμένα. για να έχουμε έτσι κάποιες απόψεις ε, ε, σε διαφορετικούς κλάδους. Επίσης ε, θέλουμε να είμαστε πιο έγκαιροι κάτι το οποίο ισχύει στην αγορά εργασίας, όχι τόσο στις άλλες έρευνες, θα αυξήσει την συγκρισιμότητα, ειδικά σαν τομέα της απασχόλησης. Θα αυξήσει επίσης την κάλυψη θεμάτων που καλύπτονται από κοινωνικά στατιστικά στοιχεία και έχουμε κατά νου το ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στο μέλλον και να προσαρμοστούμε σε μελλοντικές απαιτήσεις ε, πολιτικής. Γιατί εκεί πέρα έχουμε ένα θέμα με το ποσοστό απαντήσεων. Λοιπόν, έχω εδώ... Ε, αλφαβητικά κάποια ζητήματα που μας απασχολούν. Δεν θα τα διαβάσω όλα. Δύο σχόλια θα κάνω. Το πρώτο είναι ότι έχουμε νέα ζητήματα που εμφανίζονται για πρώτη φορά για την αναπηρία. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα έχουμε καλύτερη γνώση για μετανάστες ε, και καταγωγή το άλλο είναι ότι θα συλλέξουμε δεδομένα για την φροντίδα ηλικιωμένων και αρρώστων, τις σχετικές ανάγκες, εκπαίδευση που έχει διακοπεί, δυσκολίες στη στέγη και πληροφορίες ε, για τους άστεγους. Ε, τη μεταφορά διαγενειακή πλέον εκτιμάτων και μειονεκτημάτων, ε, ηλική στέρηση, τα οποία έχουμε πολλά νέα στοιχεία στο πλαίσιο ενό ε, καλαθιού διαφόρων δικτών, ε, ε, συνταξιοδότηση. Επίσης απασχολεί αυτό την πολιτική ποιότητα ζωής, δουλειά και οικογένεια, χρήση υπηρεσιών και υπηρεσιών φροντίδας και ανεξάρτητης αυτόνομης διαβίωσης. Διάφορα πράγματα λοιπόν που είναι καινούρια. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι το εξής. Η ομορφιά αυτών των στατιστικών στοιχείων είναι ότι μπορούμε να διασταυρώσουμε οποιοδήποτε με οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή αν μιλάμε για αναπηρία μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για την ε, αναπηρία και αγορά εργασίας. Δηλαδή τα άτομα με αναπηρία έχουν την ίδια αντιμετώπιση στην αγορά εργασίας. Ε, ή αναπηρία και εκπαίδευση, αναπηρία και εισόδημα, αναπηρία και άλλα φαινόμενα που μετράμε το ίδιο για τους μετανάστες. Ε, ένταξη μεταναστών. Ε, μετανάστες στην αγορά εργασίας, μετανάστες στην εκπαίδευση. Ε, το ίδιο για το φύλλο, την ηλικία, Να βάλουμε δηλαδή κάποια στοιχεία διακριτικής ε, μεταχείρισης ε, που μπορεί να γίνουν κάπως ε, αντικειμενικά. Αφού σας παρουσίασα λοιπόν το βασικό κορμό, έχουμε σε αυτή τη μικρή πυραμίδα όπου θα δείτε ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο τι στοιχεία συλλέγουμε και στο πώς τα συλλέγουμε τι συλλέγουμε. Δηλαδή, αυτά ορίζονται στον κανονισμό τον ίδιο, τον IESS. Ε, ε, Θα σας δείξω τις μεταβλητές και το γενικό το χάρτη σε λίγο. Ε, το πώς συλλέγουμε τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία, αυτό είναι πιο τεχνικό και αφορά εκτελεστικές πράξεις. Εδώ μιλούμε για ένα δεύτερο στρώμα, μια δεύτερη φάση δηλαδή και το αριθμό των μεταβλητών και τον τίτλο τους. Εδώ έχουμε τρεις κατεξοδότηση πράξεις ενώπιον μας. Το ένα, μία φορά το σχεδιασμό, η άλλη ε, το τίτλο των μεταβλητών ε, για την αγορά εργασίας και το τρίτο αφορά το εισόδημα και ε, τις συνθήκες διαβίωσης και έχουμε και πέντε τεχνικές εφαρμοστικές ε, πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού που έχει να κάνει με τις ποιοτικέ εκθέσεις, τεχνικά στοιχεία κοινά σε διάφορη συλλογή δεδομένων, τεχνικές λεπτομέρειες για το εργατικό δυναμικό, τεχνικές λεπτομέρειες για ε, την ε, ανεργία σε μηνιαία βάση κλπ. Πολυετής σχεδιασμός εναλλασσόμενος βασίζεται στο άρθρο 4 ε, του κανονισμού πλαίσιο. Στόχο έχει ε, να σχεδιάζει με ευελιξία τους τομείς που θα καλύπτονται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την επόμενη οκταετία κάθε φορά. Ε, στόχο έχει να ορίζει με κάποιο ευέλικτο τρόπο τη μη ετήσια συλλογή στατιστικών στοιχείων. Και ε, τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών ε, δεδομένων ε, που δεν είναι αιτήσια για την αγορά εργασίας και για τη διαβίωση. Επιλέξαμε αυτή την προσέγγιση για να μην υπάρχει ιδιαίτερο φόρτος, αλλά για να καλύπτουμε περισσότερους τομείς. Δηλαδή δεν συζητάμε, δεν ρωτάμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα ιδιαίτερα όταν είναι πιο διαρθρωτική η κατάσταση. Πιο... Ναι. Δεν είναι πάντα ίδια τα κεφάλαια που ρωτάμε. Έτσι θα μπορέσουν οι χρήστες να έχουν μια επισκόπηση, μια συνολική θεώρηση για το τι τους περιμένει και τι μπορούν να περιμένουν σε ποια χρονική στιγμή, τι, τι πληροφορίες στατιστικές μπορούν να περιμένουν και πότε. Γι' αυτό ε, θα επιτρέψει και στις Εθνικές Στατιστικές Αρχές και στη Eurostat να ε, διαχειριστούν κάπως το φόρτο και να μοιράσουν ε, το φόρτο εργασίας για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων. Τι είναι η ευελιξία αυτή που λέμε. Θέλουμε να επιμείνουμε και να τονίσουμε ότι αυτός ο κανονισμός πλαίσιο μας επιτρέπει να αναθεωρούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ε, ε, το πολυετή κυλιόμενο σχεδιασμό για να βλέπουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποια είναι τα νέα ad hoc ε, θέματα που ενδιαφέρουν τους χρήστες για να γίνεται αυτό με έναν τρόπο εύκολο στην προσαρμογή και ευέλικτο. Η δεύτερη κατεξουδότηση πράξη που έχετε ενώπιό σας είναι αυτή που αφορά ε, ε, τον αριθμό και τον τίτλο των μεταβλητών για το τομέα ε, του εργατικού δυναμικού. Είναι από τον κανονισμό αυτό τον IESS. Yes. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, τώρα στην αρχή έχουμε εντάξει μόνο το πυρήνα των θεμάτων που αφορούν την αγορά εργασίας, το εργατικό δυναμικό. Αυτό έχει να κάνει μέχρι το 2021 και τους μετανάστες και θα συμπληρωθεί προοδευτικά το 2022 όπου θα προσθέσουμε τις δεξιότητες σε αντίστοιχη κατεξοδότηση πράξη και το 2023 θα ασχοληθούμε μέχρι τα τέλη του 2023 Για το 23, ε, λοιπόν, ε, τις συντάξεις και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Year, I mean, most likely in November. Μέχρι τα τέλη του έτους, ε, κάθε φορά εννοώ περίπου το Νοέμβριο και το 22 και το 23. Η τρίτη κατεξοδότηση πράξη που έχετε μπροστά σας αφορά ε, ε την, ε, το εισόδημα και τις συνδίκες διαβίωσης. Και πάλι έχουμε ένα πολυετή κυλιόμενο σχεδιασμό. Βασικά, το 2021 έχουμε το πυρήνα και εξετάζουμε τι στοιχεία για τα παιδιά. Υγεία, στερήσεις και ε, κατάσταση των μεικτών οικογενειών ή ε, νέες οικογένειες που προκύπτουν μετά από διαζύγια. Το 2022 θα έχουμε κατεξοδότηση πράξης που θα αφορούν την υγεία, την ποιότητα ζωής και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Φέτος θα λάβετε άλλες δύο κατεξοδότηση πράξης. Η μία θα αφορά την εκπαίδευση, τη διαβίου μάθηση, την εκπαίδευση ενηλίκων. Ε, το 2022 θα γίνει αυτή η έρευνα και μια κατεξοδότηση πράξη που θα ασχολείται με τη χρήση των υπολογιστών και της τεχνολογίας πληροφορικής στα νοικοκυριά. Το 2021 όλα αυτά. Κανονικά θα λάβετε τις προτάσεις γύρω στον Ιούνιο φέτος. Αυτή ήταν η σύντομη παρουσίασή μου, αυτά τα λίγα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις από πλευράς των μελών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Μερσή για την παρουσίασή σας. Μας δώσατε στοιχεία επίσης και για την αναπηρία τα οποία έχετε συλλέξει στα πλαίσια του εργατικού δυναμικού γιατί αυτό θα βοηθήσει να εντοπίσουμε καλύτερα τις αδυναμίες που μπορεί να παρουσιάζει η αγορά. Να θυμίσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είχε πετύχει ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να υπάρχουν σε κάθε έρευνα ε, δεδομένα για την αναπηρία. Ήδη από το 2017 όταν τα Ηνωμένα Έθνη αξιολόγησαν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αναπήρων, ασκήθηκε κριτική ε, γιατί δεν ε, καταγράφουμε με τον σωστό τρόπο ε, τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρίες. Και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μια τεχνική παρατήρηση να μεταφέρεται στη Eurostat υπάρχει ακριβώς ε, με τρεις παραμέτρους ένα πλήρες πρότυπο ευρωπαϊκό το οποίο όμως, ε, από το οποίο δύο μόνο παράμετροι θα εφαρμοστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ληφθούν υπόψη καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και αναφέρεται επίσης και στο θέμα των εργαζομένων στις εξέδρες εξόριξης. I think it's, it's, it's very important for everyone to have very adequate statistical material as soon as possible. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερα στοιχεία λοιπόν και στους εργαζομένους της επιχειρήσεις του διαδικτύου, στις μεγάλες επιχειρήσεις του διαδικτύου. How, how do you have, do you have uh, foreseen to give more data on platform workers? Thank you. Thank you. Anybody else? Uh, maybe just uh, uh, Λοιπόν, οι παρατηρήσεις σας είναι ενδιαφέρουσες. Όλα αυτά που μας είπατε επίσης ε, και ε, για τα θέματα τα οποία επικαλύπτονται με πάρα πολλές προτεραιότητες ε, και προκλήσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα ακριβώς της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών. Ο κανονισμός πλαίσιο δίνει την δυνατότητα και δημιουργεί ένα πλαίσιο ε, για να ληφθούν υπόψη επιμέρους χαρακτηριστικά για τους ιδιαίτερα ευάλωτους, για τους πιο ευάλωτους ε, σε εδαφικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο με αποτελεσματικό σε επίπεδο και υπεύθυνο τρόπο έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε σωστά τους τομείς οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν τις περισσότερες ανάγκες και να μπορέσουμε να κατανείμουμε μετά τις πιστώσεις με αποτελεσματικό τρόπο. και καλό είναι που συλλέγετε ε, τα στοιχεία με τον τρόπο που το κάνετε γιατί πολλές φορές δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν οι κυβερνήσεις και μας παρέχουν με τη σειρά τους. Στην κατεξουσιοδότηση ε, πράξη Υπάρχει αναφορά επίσης περίπτωση και ε, σε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ε, στα θέματα των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων, των εργαζομένων σε ψηφιακές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα ε, για τη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων. Κύριε Μέση, έχετε ξανά το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με τις αρχικές διαστάσεις για τα ΝΑΤΣ 2, είναι σαφές ότι ε, προσπαθούμε να καλύψουμε εμείς την διαφορετικότητα σε τοπικό επίπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δώσουμε πληροφορίες οι οποίες να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη την οποία τρέφεται απέναντί μας σχετικά με τα δεδομένα τα οποία παράγουμε. Εμείς είμαστε ανεξάρτητοι, ε, νομικά ε, είμαστε ανεξάρτητοι και οι προσπάθειές μας ε, έχουν σαν στόχο το να δώσουμε πραγματικές πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία. Νομίζω ότι είναι αρκετά επιτυχές αυτό το οποίο έχει γίνει και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο κατάφερε το ίδιο το Κοινοβούλιο το οποίο επέβαλε την έρευνα για το εργατικό δυναμικό. Νομίζω ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ε, σε σχέση με την κατάσταση ε, των ανθρώπων οι οποίοι φύγονται από αναπηρίες. Το θέμα δεν είναι μόνο πληροφορίες για τις αναπηρίες, αλλά περισσότερες πληροφορίες επίσης και για άλλους τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, ε, το, το εισόδημα, ε, το ελάχιστο εισόδημα και νομίζω ότι είναι πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να συλλέξουμε, να μετατρέψουμε σε δεδομένα Δύο από τις τρεις παραμέτρους έχουν ληφθεί πλέον υπόψη από το αρχικό πρότυπο. Θα δούμε αν αυτό επαρκεί. Νομίζω ότι ε, το αρχικό πρότυπο έτσι και αλλιώς είναι ε, ε, κάτι το συνεκτικό, είναι ένα μπλοκ αλλά θα πρέπει να το ελέγξουμε. Σχετικά τώρα με τους εργαζομένους The agenda. Um, the, the, the problem there... σε σχέση με τις διαδικτυακές πλατφόρμες λοιπόν. We need to do first feasibility studies, uh, the, the, the phenomenon... Το φαινόμενο λοιπόν είναι νέο και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στον εντοπισμό αυτών, αυτού του τύπου της πλατφόρμας και των εργαζομένων που συνδέονται με τις πλατφόρμες αυτές. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν προς το παρόν είναι μια μελέτη εφικτότητα σε εισαγωγικά η οποία θα ολοκληρωθεί το 2022, θα συλλέξουμε στοιχεία παράλληλα με αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις επί τη βάση συμφωνιών κυρίων ε, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί εν πάση περιπτώσει. Οι οικονομικές δραστηριότητες ε, αυτές μας ε, απασχολούν. Προσπαθούμε λοιπόν να τα λάβουμε υπόψη μας και θα το δούμε μέσω της μελέτης αυτής των συνεπειών. Ε, θα οργανώσει η Eurostat ε, και μια διάσκεψη για το θέμα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα αυτό από πλευράς στατιστικής και είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Νομίζω ότι έχουμε και άλλη ερώτηση από την κυρία Ραφάλσκα. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ε, και θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. οργανωτικά αυτό πώς το έχετε σκεφτεί. Είστε σε επαφή με τις αρμόδιες στατιστικές αρχές, έχετε εθνικούς εμπειρογνώμονες, θα συζητάτε αυτά τα πράγματα. Ε, έχετε κάνει σχετικά βήματα, γιατί μιλάτε για τα νέα θέματα, ας πούμε, όπως είναι η μετανάστευση, τα θέματα κατοικίας, ε, ατόμων με αναπηρίες. Αυτά τα νέα θέματα είναι πολύ δύσκολα πορές φορές ε, να μετρηθούν γιατί υπάρχει δυνατότητα καν συλλογή στατιστικών στοιχείων. Το είπατε κι εσείς ο ίδιος. Θα μπορούσα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάθε 10 χρόνια γίνεται απογραφή στην Πολωνία και απογραφή και των αστέγων και έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για τους αστέγους. Εσύ πώς, εσείς πώς θέλετε να κάνετε τέτοιες στατιστικές μελέτες και να συλλέγετε στοιχεία. Κάτι άλλο που είναι δύσκολο να μετρηθεί είναι αυτές οι υπηρεσίες φροντίδας στο εσωτερικό της οικογένειας. Άλλο θέμα. Ε, θέματα μετανάστευσης. Πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί κάθε φορά θα πρέπει να δίνουμε απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνικής πολιτικής. Πώς τα μετράμε αυτά. Σήμερα έχει προχωρήσει η ψηφιοποίηση. Σε μερικά μέρη ναι. Και κανονικά είναι πιο εύκολο να συλλέγει στατιστικά στοιχεία από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι τα δεδομένα αυτά τα στατιστικά αργούν να φτάσουν σε μας. Υπάρχει μια διαφορά φάσεως. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά ε, τις υπηρεσίες φροντίδας ε, που παρέχονται στο ιστορικό μιας οικογένειας. Ας πούμε, η νεότερη γενιά φροντίζει την παλαιότερη ή αντίστροφα. Ε, we have some, Έχουμε ε, κάποια ε, κεφάλαια ad hoc που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα. Φροντίδα των παιδιών, φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι γεγονό ότι τέτοια φαινόμενα είναι πιο συχνά σε χώρες όπως είναι η Πολωνία. Και θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι θεσμοθετημένο έτσι, σε σύγκριση με άλλες χώρες ε, ναι, το λαμβάνουμε υπόψη αυτό. Για το γενικό σχόλιο. Τι κάνετε με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Να σας πω. Παραδοσιακά στη στατιστική τι κάνουμε. Προτείνουμε αυτή την νομοθεσία αποφασίζουν οι δύο συνομοθέτες, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και μετά εναπόκειται στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, την νομοθεσία και να συλλέγουν τα στατιστικά στοιχεία τους. Φυσικά πάντα συνεννοούμαστε πάνω κάτω με τα κράτη-μέλη, αλλά εκείνα είναι αυτά που μας διαβιβάζουν τις πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία. Για το θέμα των αστέγων, είναι πραγματικά σοβαρό το ζήτημα και έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης. προσπαθήσαμε με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας προς το παρόν, προσπαθήσαμε να ε, προτείνουμε μια πρώτη λύση με ερωτήσεις των συμμετεχόντων ε, στην έρευνα. Εξορισμού οι άστεγοι δεν συμμετέχουν σε τέτοιες έρευνες γιατί δεν είναι εύκολο να φτάσεις αυτούς και να τους προσεγγίσεις. Χρειάζονται άλλες μέθοδοι και άλλα μέσα. Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες γίνεται απογραφή και των αστέγων It requires very different methods. Είναι πολύ διαφορετικές οι μέθοδοι που απαιτούνται από τις στατιστικές έρευνες. Θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με διάφορες οργανώσεις, φιλανθρωπικές ενώσεις, σωματεία, για να έχουμε καταλόγους ανθρώπων που είναι άστεγοι. Μετά το πρόβλημα της έλλειψης στέγης δεν περιορίζεται σε εκείνους που ζουν στο δρόμο κυριολεκτικά. Το αντίθετο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τη δική τους στέγη και φιλοξενούνται προσωρινά ε, από φίλους, οικογένειες ε, ζουν προσωρινά σε κάποιους θεσμούς ή ιδρύματα που και αυτοί θα πρέπει να καταγράφονται όταν κάνεις μια απογραφή αστέγων. Εδώ χρειάζονται διαφορετικές μέθοδοι από τις στατιστικές έρευνες και βέβαια ο κανονισμός αυτός είναι στραμμένος περισσότερο προς τις στατιστικές έρευνες. Δεν αρνούμε τη σημασία ε, του θέματος των αστέγων, αλλά προσπαθεί να δώσει μια απάντηση και αυτό το νομοθέτημα. Τώρα για την ψηφιοποίηση προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε κατά πολύ το χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων, ιδιαίτερα από το χρόνο που έχουμε κερδίσει στην πρόσβαση των διοικητικών στατιστικών στοιχείων τουλάχιστον, θα κερδίσουμε ένα χρόνο τουλάχιστον ε, σε ό,τι αφορά τις ειδικέ διαβίωσης και το εισόδημα. Δηλαδή θα έρθουν ένα χρόνο νωρίτερα οι πληροφορίες σε σχέση με το παρελθόν με την νέα αυτή νομοθεσία. Και ενθαρρύνουμε τις εθνικές στατιστικές αρχές να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, τις νέες τεχνικές και τα νέα εργαλεία. Έχουμε κάνει μελέτες αντικτύπου για δύο έρευνες που είναι πάρα πολύ βαριές και πάρα πολύ δύσκολες για τους ε, συμμετέχοντες. Το ένα έχει να κάνει με την κατανάλωση και το άλλο έχει να κάνει με ε, την ε, χρήση του χρόνου. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα, κινητά τηλέφωνα φυσικά πάντα με την ε, συνένεση του ενδιαφερόμενου για να δούμε τι κάνει ο κόσμος στον ελεύθερο του χρόνο, ποιες είναι οι καταναλωτικές συνήθειες. Πάντα χρειάζεται η συνένεση για να γνωρίζουμε καλύτερα την καταναλωτική συμπεριφορά, τι αγοράζουν, τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους για να κερδίσουμε χρόνο. Πάντως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε με την καλή ενία το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την ανωνυμία φυσικά των στοιχείων. Αυτά από πλευρά μου. Νομίζω τελείωσα. Our side too, I think. Από δική μα πλευρά αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστώ για την παρουσίαση. Απαντήσατε σε όλε τι ερωτήσει σα. Ελπίζω να συναντηθούμε πάλι, γιατί θα χρειαστούμε τα δεδομένα μας για να μπορούμε να παίρνουμε υπεύθυνε αποφάσεις και να διαμορφώνουμε υπεύθυνε πολιτικές. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα τα πούμε αύριο σε νέα.